κρίνονται. Το πρώτο σημείο τη σημερινή διάταξη είναι δηλώσει Πρόεδρου, συγγνώμη, δηλώσει Συμβουλίου και Επιτροπή όσον αφορά το πρόγραμμα δωρεάν διανομή ειδών διατροφή. Και σχέση με αυτό τώρα να δούμε ποιο θέλει το λόγο με, με κατόπιν όσον αφορά τη διαδικασία catch the eye. Τώρα. Για το Συμβούλιο, για το σημείο σημείο διατάξης το οποίο σας ανέφερα, θα λάβει το λόγο ο κύριος Αβίσκη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εξότιμοι κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι εντάξατε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη με συνεδριάσεως διότι είναι πραγματικά πάρα πολύ βασικό στοιχείο της ε, κοινοτικής αλληλεγγύης ε, στον τη σημερινή συγκυρία. Είναι δηλαδή η ευθύνη μας έναντι των ε, φτωχότερων, των πιο αδυνάτων της κοινωνίας, εκείνων οι οποίοι ε, χωρίς να το θέλουν βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας. Οπότε σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας πω τι πρόοδος έχει σημειωθεί στο σημαντικό αυτό θέμα. Και επίσης το 2010 είναι πάρα πολύ θετικό το ότι με πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται την έκθεση Σικέρσκη τον δε Ιούλιο του 2011 ε, απευθύνεται έκκληση προς ταχεία πρόοδο στο θέμα το ώστε το πρόγραμμα να συνεχίσει να τρέχει και για το μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα για τους Ευρωπαίους. Μιλούμε για 18 εκατομμύρια οι οποίοι καλύπτονται αυτό το πρόγραμμα. Είναι άνεργοι, είναι άστιγοι, ε, μετανάστες, ηλικιωμένοι. Κόσμος που για τον ΑΒ λόγο είχαν αυτή την κακοτυχία. Ε, μιλάμε επίση και για πολυμελείς οικογένειες, μονογονοϊκές οικογένειες. Μιλάμε για 20 εκατομμύρια ανηλίκους που ζουν σε κατάσταση αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε βέβαια χιλιάδες φιλανθρωπικών ε, σωματείων που βοηθούν ε, αυτόν τον κόσμο. Έχουν πει επίση εκατοντάδε χιλιάδων εθελοντών οι οποίοι βοηθούν να δοθεί ε, φαγητό σε αυτούς. Και ναι, που μαθαίνουν να βοηθούν τους άλλους. Επί 20 χρόνια το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί και συντείνει στην υλοποίηση των στόχων της ε, κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά είναι και στόχο εδώ τη κοινωνία. Είναι θέμα κοινωνική ανάπτυξη Με αυτό το πρόγραμμα μπορούμε επίσης να πετύχουμε τους στόχους για το 2020. Έχουμε εκατομμύρια πολιτών και φιλανθρωπικών σωματείων που περιμένουν να τους δώσουμε το πράσινο φως, περιμένουν το σήμα από Στρασβούργο και Βρυξέλλες και είμαι σίγουρος ότι πολλοί μας ακούν τώρα που συζητούμε γι' αυτό. Έτσι τα αποθέματα της παρέμβασης δίνονται στον κόσμο μέσω κάποιων εγκεκριμένων οργανισμών. Και έτσι είμαστε αρρωγοί στους μη προνομιούχους της κοινωνίας μας. Είχαμε επίσης κάποιες αλλαγές στην κοινωνική πολιτική, τελευταία. Οπότε πλέον δεν έχουμε αυτού του είδους την, την ξαγορά, η αγορά προϊόντων μέσω της παρέμβασης. Δεν ισχύει αυτό της οργανώσει αγοράς ή είναι πολύ περιορισμένο για κάποιου κλάδου για κάποια αγροτικά προϊόντα. Ε, και επίση πάρα πολλά τρόφιμα αγοράστηκαν από την αγορά για να χρησιμοποιηθούν για το πρόγραμμα. ελοχεύτερο, κάποιος κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι τα αποθέματα το 2013 να είναι ακόμα λιγότερα από το 2012. Οπότε θα πρέπει εδώ για τώρα να σας βεβαιώσω πώς θα θέλαμε να δεσμευτούμε όσον αφορά τη συνέχιση αυτού του στο Συμβούλιο τα περισσότερα κρατημέλη είπαν το ναι. Όμω υπάρχει μια παρεμποδίουσα μειοψηφία. Έχουμε κάποιε χώρε οι οποίε θέλουν να βάλουν φραγμό στη συνέχιση του προγράμματο και χρησιμοποιούν για να προτάξουν τι θέσει του διάφορα επιχειρήματα, οι περισσότεροι εξ αυτών αναφέρουν ότι πρόκειται για πρόγραμμα κοινωνική πολιτική. Η κοινωνική πολιτική θα πρέπει να είναι στα χέρια των κρατών μελών. Είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να βοηθεί τους αδυνάτους από τον κοινωνικό προϋπολογισμό. Ε, πάρα πολύ δύσκολο να χωνέψει κανείς τέτοια επιχειρήματα. Ε, δεν είναι ο ρόλος μας να κατακρίνουμε και να επικρίνουμε αυτά τα κράτη-μέλη, αλλά αλληλεγγύη θα πει να βοηθεί κανείς αυτούς που περισσότερο χρειάζονται βοήθεια. Και βέβαια η συμμετοχή στο πρόγραμμα έτσι για αλλιώς όπως ξέρουμε είναι ε, εθελοντική. Έχουμε 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως που από τον κοινωνικό προπολογισμό. Το πρόγραμμα αυτό κοστίζει ε, μόλις μεταβίας ένα ευρώ στον κάθε Ευρωπαίο πολίτη και το είπε τον Απρίλιο του 2010 ο, ο Επίτροπος ότι δεν υπάρχει κανένα φραγμό το συνεληφθεί η πολιτική για το πρόγραμμα. Για πέντε μήνε μετά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα τροποποιημένο νομοθετικό κείμενο και αν εγκριθεί αυτό το κείμενο θα λυθεί το θέμα της αγοράς των προϊόντων από την αγορά. Επομένως, τώρα το μπαλάκι είναι στο κήπεδο του Κοινοβουλίου και δεν υπάρχουν νομικοί λόγοι ε, που να τους χρησιμοποιούμε ως πρόφαση για να μην συνεχίζεται αυτό το πρόγραμμα. Επομένω, γι' αυτό σα λέω ότι απόκειται σε κάποια κράτη το, το να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό. Και εάν σταματήσει το, πρόγραμμα, το πρόγραμμα δεν θα κρυζώσουμε τη φτώχεια. Γιατί πρόκειται βεβαίως σαν να είναι κάποιος άρρωστος και απλά να, να σπάει το θερμόμετρο. Αρνείται την ύπαρξη προβλήματος. Όπως ξέρετε, ε, η Κομισιόν έχει προτείνει να περάσει η χρηματοδότηση του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων από τον τίτλο 1 στον τίτλο 2. Ο πρόγραμμα εντάσσεται καλύτερα στη στρατηγική του 2020. Η Κομισιόν θα υποβάλει μια νέα νομοθετική πρόταση για την περίοδο μετά το 2014. Ελπίζω το πρόγραμμα τότε να το υποστηρίξουν όλα τα κράτη-μέλη. Βεβαίως, η φτώχεια δεν θα εξαλειφθεί μόνο με το πρόγραμμα αυτό, αλλά μπορεί να βοηθήσει να μειωθεί η φτώχεια. Ακόμα και στα πλουσιότερα κράτη-μέλη υπάρχουν άνθρωποι φτωχοί και βεβαίω η φτώχεια δεν επηρεάζει μόνο τις μεγάλες πόλεις, αλλά και τις μικρές πόλεις και αεροκατοικημένε περιοχές υπέδρου. Και πέρα οι πιο φτωχοί άνθρωποι. Καθώς αυξάνεται η ανεργία, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Κάποιος πρέπει να τους βοηθήσει και θα έπρεπε να τους βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και το θέμα αυτό στο Συμβούλιο Γεωργίας του Σεπτεμβρίου. Κατόπιν πρωτοβουλίας της Πολωνικής Προεδρίας έλαβε χώρα μια δημόσια συζήτηση η οποία μεταδόθηκε από το διαδίκτυο. Δυστυχώς για τρία χρόνια είχαμε αδιέξοδο στο Συμβούλιο και είναι κρίμα σε μια εποχή που υπάρχει κρίση και ο κόσμος κυριολεκτικά χρειάζεται αυτή η βοήθεια, κάποιοι πολιτικοί δεν έχουν την παραμικρή αίσθηση ανθρώπινης αλληλεγγύης. Το θέμα της δωρεάν διανομής τροφίμων θα συζητηθεί πιθανότατα στην διάσκεψη Υπουργών Κοινωνικής Πρόνοιας του Οκτωβρίου. Σας διαβεβαιώ λοιπόν πω η Προεδρία κάνει ό,τι μπορεί για να βρει μια λύση στο πλαίσιο των υφιστάμενων διμερών επαφών με τα κράτη-μέλη τα οποία είναι κατά της πρότασης. Πρόκειται για επαφές μεταξύ Υπουργών Γεωργίας και Πρωθυπουργών. Ξέρω πως κάποιες αντιπροσωπείε. σκέφτονται πως το ζήτημα αυτό θα πρέπει να είναι στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 17 και 18 Οκτωβρίου και θα απευθύνουμε επιστολή στον πρόεδρο Φαν Ρόμπαϊ με αυτό το περιεχόμενο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Προεδρία γνωρίζει την στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις προτάσεις της Κομισιόν. Πολλά κράτη-μέλη επίσης στηρίζουν αυτές τις προτάσεις. Σας διαβεβαιώ πως θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να έχουμε μια θετική θέση του Συμβουλίου. Οι τελευταίες πέντε προεδρίες δεν ήταν σε θέση να ε, άρουν το αδιέξοδο. Αλλά πιστεύω πως ε, με την πολωνική ηγεσία θα τα καταφέρουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και τους βουλευτές για τη στήριξή τους στο πρόγραμμα, αλλά απευθύνομαι σε εσά με μία έκκληση να πιέσετε τις κυβερνήσεις σας και τους συναδέλφους σας βουλευτές που για τον χύψη λόγο αντιτίθενται στη δωρεάν διανομή τροφίμων πιο αδύναμους. Το πρόγραμμα αυτό αντικατοπτρίζει την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την αίσθηση ευθύνη που έχουμε για τα ασθενέστερα μέλη τη κοινωνία μας. Προωθεί τα ιδανικά μας. Υπάρχουν εκατομμύρια πολιτών της Ένωση που γνωρίζουν πως σε έναν καιρό δύσκολο δεν θα τους παραμελήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ να φανταστώ να σταματήσει αυτή τη στιγμή αυτό το πρόγραμμα. Είναι άσχημο όχι μόνο για την εικόνα της Ένωσης, αλλά όλοι μαζί νομίζω θα χάσουμε. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα για την Κομισιόν έχει ο κύριος Σιόλος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό και επικαιρότητα ε, το θέμα της ε, δωρεάν διανομής τροφίμων ε, στους φτωχούς. Μετά από τη σημαντική οικονομική κρίση, ο αριθμός των πολιτών που ζητούν τη βοήθεια αυτού του προγράμματος μπορεί να αυξηθεί δραματικά. Οι ουρές μπροστά από τις φιλοτροπικές οργανώσεις το καταμαρτυρούν. Εδώ και 25 χρόνια εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα που έχει αποδείξει την αξία του στηρίζοντας αυτές τις οργανώσεις. 440 ε, εκατομμύρια τόνοι ε, χιλιάδες τόνοι μάλλον έχουν δοθεί ε, κάθε φορά, ε, κάθε χρόνο και 18 εκατομμύρια άνθρωποι είναι οι δικαιούχοι αυτού του προγράμματος κατά μέσο όρο ετησίως. το πρόγραμμα αυτό υπάρχει και λειτουργεί σωστά και ορισμένοι θέλουν να το εξαλείψουν ακριβώς αυτή τη στιγμή που το έχουμε περισσότερο ανάγκη. Και εγώ θα είμαι πολύ σαφής για αυτή το τομέα. Οι νομικές πτυχές και οι οικονομικές πτυχές για να μπορέσει να συνεχιστεί το πρόγραμμα όραμα μπορούν να επιληθούν για την περίοδο 2012 και για το 2013. Αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση και σε αυτό θα πρέπει να είμαι σαφής. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από ένα, μια απόφαση του ΔΕΚ. Η απόφαση του ΔΕΚ δεν αμφισβητεί τη σκοπιμότητα αυτού του προγράμματος. Αυτό που αμφισβητεί είναι η νομική του βάση που πρέπει να ενημερωθεί και ακριβώ τα πολιτικά όργανα είναι αυτά που θα πρέπει να αποφασίσουν για την αλλαγή τη νομική βάση. Από αυτή την άποψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σαφώ ε, προβεί στην επιλογή τη γιατί για την περίοδο μετά το 2013 έχει ήδη προτείνει στο πλαίσιο των προτάσεών τη για το νέο ε, πολιετέ ε, χρηματοοικονομικό πλαίσιο να εντάξει το πρόγραμμα στην πολιτική οικονομική και κοινωνική συνοχή με 5,5 ευρώ για την περίοδο 2014 μέχρι 2020, ακριβώς έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η διάρκεια αυτού του προγράμματος. Για το 2012 και 2013 που συζητάμε τώρα και που αποτελούν και την επίγου, το, επίγον θέμα, η Κομισιόν και το Συμβούλιο έχουν αρχίσει να συζητούν από το 2008 ε, και το τροποποιήσαμε το 2010 για να λάβουμε υπόψη τις δικές σας παρατηρήσεις, πράγμα το οποίο θα επέτρεπε να γίνει η σύνδεση μεταξύ του σημερινού κανονισμού και το 2014 από την από το οποίο θα έχουμε νέα νομική βάση στο πλαίσιο της ε, πολιτικής κοινωνικής συνοχής. Έχω ήδη προειδοποιήσει το Συμβούλιο, όπως το είπε και ο Προεδρεύων Σαβίσκη, ότι αν δεν ληφθεί τέτοια απόφαση από πλευρά του Συμβουλίου τώρα, γιατί το Κοινοβούλιο ήδη έχει εκφράσει τη θέση του, το πρόγραμμα του 2012 δεν θα αποτελείται από το 1, παρά μόνο από το 1 τέταρτο των περασμένων ετών και για το 2013 δεν θα υπάρξει πρόγραμμα τέτοιο. Γιατί είναι κάπως απίθανο να γίνει παρέμβαση στην αγορά για να χρησιμοποιήσουμε σε σημαντικό βαθμό τις δημόσιες δημόσιες, ε, τα δημόσια αποθέματα. Άρα λοιπόν αν δεν ληφθεί αυτή η πολιτική φύση απόφαση δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε ούτε ένα ευρώ για το 2013 ενώ υπάρχει το κονδύλι. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να σας ευχαριστήσω για την μόνιμη υποστήριξή σας για αυτό το θέμα και κυρίως για το πρόσφατο ψήφισμα της 7ης Ιουλίου που τονίζει την ανάγκη εξέβρεσης μιας συμφωνίας που θα επιτρέψει τη συνέχιση αυτής, ε, αυτού του προγράμματος. Γνωρίζω επίσης πως πολλοί από εσά εξέφρασαν την επιθυμία στο να συνεχίσει η χρηματοδότηση του προγράμματος ε, στο σύνολό του από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και ως προς αυτό εγώ εξέφρασα την ευελιξία μου για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε όλα τα κράτη-μέλη που ενδιαφέρονται να μπορούν να συμμετέχουν. Και το είπα και στο Συμβούλιο ότι είμαι έτοιμο να δείξω αυτή την ευελιξία εάν το Συμβούλιο καταφέρει να βρει μια πλειοψηφία για να ληφθεί η σχετική απόφαση. Σημείωσα την συζήτηση που έγινε στο Συμβούλιο στις 20 Σεπτεμβρίου και η Κομισιόν εξετάζει αυτή τη στιγμή τις εναλλακτικές λύσεις ώστε να προσπαθήσει να επιμπλέξει την κατάσταση και ενδεχομένως να προτείνει μια κοινή νομική βάση για την κοινή γεωργική πολιτική και την κοινωνική πολιτική από τώρα ώστε για τα επόμενα έτη 2012 και 2013 να έχουμε ήδη αυτή την κοινή νομική βάση. Και ελπίζω πως έτσι θα απεμπλακεί η πολιτική κατάσταση στο πλαίσιο του ε, Συμβουλίου. Βασίζομαι στη δική σας δραστήρια στήριξη ώστε να καταστεί δυνατή μια γρήγορη συμφωνία, καθώς πιστεύω πως πρόκειται για μια επιπλέον ευκαιρία ώστε να δείξουμε πως η Ευρώπη δεν σημαίνει μόνο Βρυξέλλες και Στρασβούργο, αλλά ότι η Ευρώπη είναι, ε, βρίσκεται τόπου ε, και επειδή αυτό το πρόγραμμα υλοποιείται επί τόπου δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να την ε, αναλάβουμε ε, δηλαδή να συγκεκριμενοποιείται έτσι το ιδανικό μας αυτή η αρχή και κάθε συγκεκριμένο πρόγραμμα που φτάνει στους πολίτες και δείχνει την αλληλεγγύη που υπάρχει. Σας ευχαριστούμε Επίτροπε. Θα μπούμε τώρα, θα ακούσουμε τους ομιλητές που παρεμβαίνουν ως εκπρόσωποι των ομάδων τους και καταρχήν το λόγο θα έχει ο κύριος Σικέρσκι εξ ονόματος του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίε και κύριοι. Η κρίση σοβεί εδώ και αρκετό καιρό. Ανθρώπινες ζωές συνεχώς γίνονται λένε και πιο αφόρητες μειώνονται οι μισθοί, χάνονται θέσει εργασία, ε, ε, αυξάνονται οι τιμέ των τροφίμων και ο κόσμο θα πρέπει όμω να ε, αγοράσει ας πούμε, τα φάρμακα για τυχόν ασθένειε και δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν τρόφιμα. Επομένω, πιάνει τόπο αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε 80 εκατομμύρια οι οποίοι ζουν κάτω από το από τη φτώχεια και εκεί γύρω. Οπότε δεν είναι δυνατόν να πούμε σε αυτόν τον κόσμο ότι θα, θα κλείσει βρίσκα, θα, θα κοπούν αυτά τα χρήματα για τα δωρεάν τρόφιμα. Η παρέμβαση και οι σχετικές ε, αγορές προϊόντων έχουν συρρυκνωθεί πάρα πολύ. Οπότε θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε, πώς θα μπορέσουμε να διαθέσουμε αυτά τα τρόφιμα στον κόσμο που τα χρειάζεται. Εδώ, σε αυτό το κοινοβούλιο, έχει συζητηθεί το θέμα και ε, σχεδόν ομόφωνα είπαμε το ναι. Ε, θα πρέπει να συνεχιστεί να τρέχει αυτό το πρόγραμμα ακριβώς όπως και στα επίπεδα που κινείται τώρα. Ε, πολλές εκλογές έχουμε προέλθει και δεν ξέρω τι γίνεται γιατί πολλές φορές λένε τα δεσμικά όργανα για αλληλεγγύη οπότε υπάρχει κάποια αντίφαση. Η καταπληκτική της φτώχειας είναι και ένας από τους στόχους της στρατηγική για το 2020. Βέβαια, κρίνουμε πάρα πολύ θετικό το ότι ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ε, στην ομιλία του σήμερα το πρωί το πόσο σημαντικό πρόγραμμα είναι αυτό. Οπότε θα πρέπει να πούμε στου συναδέλφου από τι χώρε που βάζουν φραγμό σε αυτό το πρόγραμμα ότι θα πρέπει να μεταβάλουν τι απόψει του. Στην περίοδο του 2014 μέχρι 2020 έχουμε τα 250 εκατομμύρια ετησίω τα οποία έχουν διατεθεί για το πρόγραμμα. Μέχρι τώρα έχουμε 500. Άρα αυτό πάει να πει περικοπή 33%. Άρα θα πρέπει να φτάσουμε στα, στα, στα 3,5 δις όπως θέλουμε. Και τώρα, ο κύριος Καπούλας Άντος είναι ο επόμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση που κάνουμε σήμερα δεν θα έπρεπε καν να γίνεται κοινή λογική και το αίσθημα της αλληλεγγύης θα έπρεπε ήδη να έχουν λύσει το πρόβλημα που σήμερα συζητάμε. Στον ευρωπαϊκό χώρο που θεωρούμε ότι είναι το λίκνο της ευημερία, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης υπάρχουν σήμερα σύμφωνα με τους ίδιους τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω από 40 εκατομμύρια άνθρωποι που κινδυνεύουν από ε, φτώχεια όσον αφορά τα τρόφιμα έχουν ε, διανεμηθεί σε 440.000 τόνοι σε κόσμο. Κανείς δεν αφιβάλλει ότι το 2012 η κατάσταση θα είναι χειρότερη. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που δεν πάβει να βαθαίνει θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο κόσμο και οικογένειες σε ένα πλαίσιο στο οποίο οι κοινωνικές πολιτικές έχουν περικοπεί κατά σε μεγάλο βαθμό. Είναι λοιπόν ακατανόητη και απαράδεκτη η στάση 6 των μελών που μπλοκάρουν την νομική βάση ώστε να μπορέσει να διατηρηθεί η διανομή τροφίμων, η επιστημιστική βοήθεια για το 2012 και 2013. Εγώ χαιρετίζω αντιθέτω την χειρονομία της Κομισιόν στο, άτομο του κυρίου Επιτρόπου που κάνει ό,τι μπορεί για να ε, παρακάμψει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μέσω της απόφασης του 10. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δείχνει κοινωνική αναισθησία που είναι αντίθετη στις αξίες μας και στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Η θέση του Υπουργού, του Υπουργείου Γεωργίας και της Πολωνίας, του αρχηγού της Πολωνίας και του Υπουργού Γεωργίας της θα πρέπει να μπορέσει να επιλύσει διαμιάς πια αυτό το πρόβλημα έτσι ώστε να απαντήσουμε με αλληλεγγύη και δικαιοσύνη που είναι το, τα εμβλήματα της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Λουίς και τώρα εξ ονόματος των φιλελευθέρων για δύο λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Τζόρτζ Λάιον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ. Βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση σήμερα όσον αφορά αυτό το πρόγραμμα. Κατά την άποψή μου, δεν θέλω να το καταστήσω σαφές, πιστεύω πως το πρόγραμμα αυτό είναι ζήτημα κοινωνικής πολιτικής και όχι γεωργικής πολιτικής και θεωρώ πως θα έπρεπε να προχωρήσουμε παραπέρα και να είναι εθνική ευθύνη. Γι' αυτό υποστηρίζουμε αυτό το οποίο προτείνει η Κομισιόν για το πολιετές μουσιονομικό πλαίσιο του 2014 και ανοίγει το δρόμο να μετακινηθεί από τον τίτλο 1 στον τίτλο 2. Όμως η κατάσταση σημερινή όσον αφορά τα επόμενα δύο έτη του προγράμματος είναι εντελώς απαράδεκτη. Πρέπει να βρεθεί μια γρήγορη λύση. Ο κίνδυνος είναι σαφής. Τα χρήματα τα οποία διατίθενται σε φιλανθρωπικές οργανώσεις σε 20 κράτες θα πάνε από 500 στα 100 εκατομμύρια ευρώ και το Συμβούλιο συνεχίζει να μπλοκάρει τη λύση και αφήνει 18 εκατομμύρια ανθρώπους στην μοίρα τους. Αυτή είναι η σκανδαλώδης κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Δεν είναι δυνατόν στην Ευρώπη του 21ου αιώνα και ειδικά σε καιρό κρίσης. Πρέπει να αφήσουμε το Συμβούλιο να, αναλάβει να πάρει στα σοβαρά τις ευθύνες του. Ανεξαρτήτως του αν το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι εθνικό ή κοινωνική πολιτική, πρέπει να βρεθεί ένα τρόπο να λυθεί αυτό το πρόβλημα για τα επόμενα δύο χρόνια. Θα βρεθεί μια μεταβατική λύση για τα επόμενα δύο έτη και το Συμβούλιο θα συνεργαστεί με Κομισιόν και Κοινοβούλιο για να λυθεί το ζήτημα. Πρέπει να βρεθεί μια λύση βραχυπρόθεσμη και είναι απαράδεκτο οι φτωχότεροι να καθίστανται όμοιροι αυτής της διαμάχης και της αδυναμίας του Συμβουλίου να βρει μια κοινή γραμμή. Πρέπει τώρα οι Εθνικέ κυβερνήσει να πάρουν στα σοβαρά τι ευθύνε του και να συνεργαστούν με την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο για να βρούμε γρήγορη λύση έτσι ώστε όσοι χρειάζονται αυτό το πρόγραμμα το 2012 και 2013 να μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν. Ευχαριστώ κύριε Λάιον για τους συντηρητικού και μεταρρυθμιστές για 1,5 λεπτό ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ όπως και ο τελευταίος ομιλητής, νομίζω και εγώ πως είμαστε σε δύσκολη θέση όσον αφορά αυτό το θέμα. Αναγνωρίζω βεβαίως πως έχουν βοηθεί πάνω από 18 εκατομμύρια άνθρωποι. Έχει κάνει φοβερή δουλειά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα είμαστε σε θέση αμφισβήτησης της χρηματοδότησης και οφείλω να πω πως πρέπει να το δούμε αυτό το ζήτημα το είπε ο κύριο Υπουργός πως τα αποθέματα του 2013 θα είναι πιο περιορισμένα από του 2012. Και αυτή είναι η πραγματικότητα γιατί όλοι γνωρίζουμε πως η ασφάλεια τροφίμων δεν είναι αυτή που ήταν στο παρελθόν και αυτό αποτελούσε φοβερή πρόκληση για όλου μα. Αλλά θα ήθελα να πω το εξή. Δεν ξέρω εάν αυτό πρέπει να έρθει από τον προπολογισμό, το γεωργικό ή τον κοινωνικό. Πρέπει να το πετύχουμε σωστά. Δεν μπορούμε απλά να αυτοσχεδιάσουμε επειδή δεν διαφωνούμε με κάτι. Οπότε, ποιο ταμείο θα πληρώσει. Αυτή είναι η ουσία εδώ πέρα. Και θα ζητούσα τον κύριο Τσόλος, θα ρωτούσα τον κύριο Τσόλο το εξή. Είναι αποτελεσματική αυτή η πολιτική. Όλοι γνωρίζουμε για τις σπατάλη τροφίμων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι αυτός ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια. Αντιλαμβάνουμε λοιπόν πως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος φτώχεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αναγνωρίζω αυτό και να βοηθήσουμε, αλλά ελπίζω ειλικρινά να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα αυτό και θέλω να τη βρει τη λύση αυτή το Συμβούλιο Γεωργίας γιατί δεν πιστεύω πως μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια αλλά δεν πιστεύω πως αντιμετωπίζουμε σωστά το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Για τώρα για λεπτά το λόγο έχει η κυρία Καρίμα Ντελή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ. Ο αριθμός των ανηρών και των φτωχών αυξάνεται. 43 εκατομμύρια και πάνω απειλούνται από έλλειψη τροφίμων. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Έξι κράτη-μέλη όμω θέλουν να βάλουν τα φόρμακα στο πρόγραμμα χωρί να προτείνουν κάποια εναλλακτική. Γερμανία, Σουηδία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτω χώρε και η Τσεχική Δημοκρατία. Βεβαίω ε, υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου θα πρέπει να την τηρήσουμε. Οπότε είχαμε αποφανθεί τον Ιούλιο με πρωτοβουλία των Πρασίνων. Είχαν γίνει οι πρόεδρε πάρα πολύ εύστοχε προτάσει για να σωθεί το πρόγραμμα. Οι πράσινοι προτίθεται να συνεργαστούν μαζί σα και να βρεθεί μια μακρόπνοη λύση. Άπαξ όμω και έχουμε εκατομμύρια που εξαρτωθώ το πρόγραμμα. Δεν είναι δυνατόν να, να, να υποτετραπλασιάσουμε την πρικοδότηση. Επομένω το πρόβλημα είναι πραγματικό. Αν δεν γίνει κάτι μέχρι τώρα θα, θα λείψουν αυτά τα 300 εκατομμύρια και τίποτα δεν εγγυάται το ότι θα μπορέσουν οι εθνικέ κυβερνήσει να αντισταθμίσουν ε, αυτή την έλλειψη. Είναι θέμα ουσιαστικό, είναι θέμα ελληνίδα των λαών. Να μην αφήσουμε μια μειοψηφία ανεύθυνη των ε, κυβερνήσεων να στήσουν τα τρόφιμα αυτά του Ευρωπαίου. Γιατί είναι θέμα επιβίωση. Η καταπολέμηση τη φτώχεια και η κακή διατροφή δεν είναι θέμα μόνο κάποια μεταρρύθμιση τη. Θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπο παραγωγή και να μπορέσουμε η παραγωγή των τροφίμων να είναι πιο κοντά στον κόσμο ε, και κυρίω ε, πιο κοντά στους φτωχότερους οι οποίοι και αυτοί έχουν δικαίωμα σε μια υγιεινή διατροφή και έτσι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το να ε, λείπουν τα τρόφιμα από όλο ένα και λιγότερους. Οπότε θα πρέπει αυτοί ε, που χρειάζονται να μπορέσουν να προσφύγουν σε αυτή τη λύση. Θα πρέπει οι επόμενες ε, προεδρίες από τον Ιανουάριο και πέρα να μπορούσαν να επανεξαφέρουν τη λογική στο Συμβούλιο. Γιατί θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι είναι ε, λογική ανάγκη είναι, είναι επιτακτική ανάγκη. Όταν για τις τράπεζες βρίσκεται λύση, σώζεται τις τράπεζες, αλλά όταν, για τους ανθρώπους όχι. Τα είπαμε τελευταία φορά. Τα ανθρώπινα όντα είναι πιο σημαντικά από τα χρηματιστήρια, από τα χρηματοοικονομικά. Ήρθε η ώρα να το ε, ασπαστούμε αυτό, να το καταλάβουμε. Θα πρέπει μένως να ανανεώσουμε αυτή μας την προσπάθεια με τρόπο επικοδομητικό. Σε ευχαριστώ κυρία συνάδελφο, ο πρόεδρος και τώρα για την Ευρωπαϊκή Νοτική Αριστερά έχει το λόγο για ένα λεπτό η κυρία Καβιτσίνα. Οι άνθρωποι που υποφέρουν δεν αξίζουν λύπηση ή κινησμό, αλλά βοήθεια. Χθε εδώ μέσα συζητούσαμε για τις αμψόμενες χώρες και την διατροφική ασφάλεια και σήμερα βλέπουμε το ότι κάποιες κυβερνήσεις όπως η Γερμανία, Δανία, Τσεχία, Σουηδία, Ολλανδία και Μεγάλη Βρετανία εσκεμένα περιορίζουν δικαιώματα αυτών των ανθρώπων με το να μην επιτρέπουν να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα. 43 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση απειλούνται από αυτό το ζήτημα, δηλαδή μία μέρα στις δύο μπορούν να τραφούν πλήρως. 19 εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται πλήρως από αυτό το πρόγραμμα. Το 2010 ήταν το ευρωπαϊκό έτος κατά της φτώχειας. Με διάφορα εκεί πέρα συνθήματα. Όποιος θεωρεί τη φτώχεια μόνο αριθμούς, καλό είναι να σκεφτεί πως θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους ώστε τουλάχιστον να έχουν τα απολύτως βασικά. Σας ευχαριστώ για τους μη εγγεγραμμένους. Ο κύριος Στογιάνοφ, 1,5 λεπτό. Το πρώτο το οποίο έμαθα στο Πανεπιστήμιο ήταν ότι τίποτα δεν είναι τζάμπα στη ζωή. Έχουμε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων στη χώρα μας παίρνουν 150 ευρώ σύνταξη και αφού αγοράσουν τα φάρμακά του και τι βασικέ υπηρεσίε, δεν του μένουν χρήματα για να μπορούν να πάρουν, να αγοράσουν φαγητό. Κύριε Σαββίτσκι, είπατε ότι πρέπει να πληρώσουμε ο καθένα ένα ευρώ για τη χρηματοδότηση του προγράμματο. Αλλά αυτοί οι συνταξιούχοι στη Βουλγαρία έχουν εισφέρει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το πρόγραμμα. Δεν λειτουργεί στη Βουλγαρία το πρόγραμμα αυτό δεν αποδίδει. Δηλαδή. Να συνεχίσει να τρέχει το πρόγραμμα. Αλλά κύριε Επίτροπε, και εσείς και η Επιτροπή να κάνετε ό,τι πρέπει ούτω ώστε να είναι προσβάσιμο αυτό το πρόγραμμα. Αλλά για όλους τους Ευρωπαίους και όλα τα κράτη-μέλη. Κύριε Τζίμερ, επίσης σας ευχαριστούμε που είπατε αυτά που είπατε για τις χώρες που δεν εγκρίνουν το πρόγραμμα. να τους κατονομάσουμε. Όλοι σήμερα μας ακούνε να ξέρουν ποιοι είναι εκείνοι που βάζουν φραγμό στην διανομή των δωρεάν τροφίμων. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα τελείωσε ο κύριος των αγορεύσεων για ε, τις πολιτικές ομάδες και τώρα πάμε στους ε, κατάτομων ε, αγορητές. Για δύο λεπτά πρώτος ο κύριος Άλμπερτ Ντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Επίτροπε και κύριε Υπουργέ, πολλά κράτη-μέλη και πολλοί συνάδελφοι ήταν υπέρ της συνέχισης αυτού του προγράμματος και γι' αυτό όπως ακούσαμε ε, χρειάζεται η συνέχιση αυτού του προγράμματος. Όμως αυτό είναι κυρίως αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι στην Ευρώπη που δεν έχουν να φάνε. Είναι ευθύνη των κρατών μελών να το φροντίσουν αυτό. Στη Γερμανία υπάρχουν νόμοι που εγγυούνται την διατροφή για όλους τους Γερμανούς πολίτες. Η απόφαση του ΔΕΚ άλλαξε το υπάρχον πλαίσιο. Ορίστηκαν συγκεκριμένα όρια. Το δικαστήριο διαπίστωσε πως το τρέχον πρόγραμμα υπό τη μορφή του δεν είναι συμβατό με την συνθήκη. Γνωρίζω πως πρέπει να βρεθούν απαντήσεις για να συνεχιστεί η βοήθεια για εκατομμύρια ανθρώπων που την έχουν ανάγκη, αλλά τονίζω ακόμη μία φορά. Η ευθύνη για την κοινωνική πολιτική είναι των κρατών μελών. Ίσως θα έπρεπε να το σκεφτούμε. Μήπως θα ήταν καλύτερο αντί για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα να έχουμε προγράμματα των κρατών μελών τα οποία θα μπορούσαν να συγχρηματοδοτηθούν από εμάς για να διασφαλιστεί η επάρκεια τροφίμων σε όλα τα κράτη-μέλη. Για να υπάρχει και μη διασφάλιση και να συνεχιστούν τα προγράμματα. Η ομάδα του ΕΛΚΟ οπωσδήποτε θα συνεργαστεί για να βρεθούν λύσεις. Το έζησα στη Βραζιλία κάποτε που είχα πάει το πώς μας ζητούσαν οι Βραζιλιάνοι τα αποφάγια μας. Ήταν σοκ σε μια τόσο πλούσια γεωργική χώρα να ζω αυτό το πράγμα και δεν θα πρέπει να γίνει στην Ευρώπη να μην έχει ο κόσμος να φάει. Σας ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό, το Δεκάστρο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Μάρε Ξαβίνσκε, αγαπητέ Επίτροπε Ντάσιαν Τσόλο, το πρόγραμμα δωρεάν διανομή τροφίμων στου πολίτε που κινδυνεύουν από φτώχεια αντιπροσωπεύει ένα πολύ σημαντικό μέσο για την βοήθεια προ τι πιο αδύναμε τάξει τη κοινωνία μα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει χαρακτηρίσει την επιτυχία τη γεωργική ε, πολιτική των τελευταίων ετών και που επιτρέπει 440.000 ε, τόνοι τροφίμων να διανέμονται ετησίω σε ένα σωρό οικογένειε και ανθρώπους που δυσκολεύονται. Και ο αριθμός των φτωχών θα αυξηθεί τη στιγμή που ε, το δικαίωμα πρόσβαση στα τρόφιμα θεωρείται πλέον ένα θεμελιώδες δικαίωμα, ανθρώπινο δικαίωμα. Και αυτό δεν μπορεί να μπλοκάρεται μόνο και μόνο από του υπουργού Γεωργίων. Γνωρίζουμε την απόφαση του 10 και θα εργαστούμε ώστε να υπάρξει κείμενο μετά το 2013 που να λαμβάνει υπόψη τα παρατηρήσει του 10. Ωστόσο δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να διακοπεί αυτό το πρόγραμμα. Πιστεύω ότι ενώ η Ευρώπη σήμερα συζητά για 500 εκατομμύρια ευρώ για βοήθεια στους πολίτες της, ΗΠΑ, ο Αμερικανικός νόμος το Farm βοηθά τους πολίτες του με πάνω από 20 δις ε, δολάρια. Είναι λοιπόν απαραίτητο να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και ευχαριστώ με την ευκαιρία τον Υπουργό Σαββίσκη και την Πολωνική Προεδρία και το θάρρος και την ε, δύναμη με την οποία ο Επίτροπος ε, υποστηρίζει αυτή την υπόθεση. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Πάολο. Ε, τώρα έχει το λόγο για 1,5 λεπτό ο κύριος Έλγουαρντ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 43 εκατομμύρια σήμερα βρίσκονται σε κατάσταση και δεν μπορούν να βρουν φαγητά. Να υπάρχει μέρα παραμέρα θα έπρεπε κάποιο κοτόπουλο ψάρι θα πρέπει τώρα να σταματήσουμε αυτή την, την τάση που με λόγους γραφειοκρατικούς θέλουν να μπλοκάρουν αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε στόχους για το 2020 μεταξύ των οποίων είναι και ο κοινωνικός αποκλεισμός να σταματήσει αλλά και η φτώχεια και αυτό το πρόγραμμα αυτό κάνει εξυπηρετή και έχει άμεσα αποτελέσματα. Όμω θα πρέπει να δούμε τι ε, πραγματικέ αιτίε τη φτώχεια, αλλά από την άλλη μεριά να καλύψουμε και αυτού που δεν έχουν χρήματα να μπορέσουν να θρέψουν αυτού και την οικογένειά του. Έχουμε πάρα πολλά προγράμματα που βοηθάνε τους φτωχού και την κοινωνικό αποκλεισμό. Ε, πολλές φορές αυτά όμως μένουν νεκρό γράμμα και δεν ωφελούνται οι πολίτες. Και σε 19 κρατημέλη έχουμε 30 ε, εκατομμύρια οι οποίοι ωφελούνται από τις φιλοδομικά σωματεία και επομένως ε, επιτόπου δίνεται βοήθεια σε αυτούς που τη χρειάζονται περισσότερο. Κάποια λογική, αν όχι, το να συμπάσχει κανείς απαιτείται από τους ε, ηγέτες των χώρων. Ευχαριστούμε το Συμβούλιο για το όσα είπε, αλλά και τον Επίτροπο. Δεν είναι τώρα ε, ώρα κανείς να παίζει παιχνίδια μικροπολιτικά με ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε κύριε Έλγορτ για ένα λεπτό τώρα έχει το λόγο κυρία Ήλτα Φιγκερέντα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήδη επανειλημμένως έχουμε υπογραμμίσει εδώ τη σημασία διατήρησης ενός προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων από τη στιγμή που έχουμε 18 εκατομμύρια ανθρώπους όπως το 2009 και μάλιστα εκατομμύρια ανθρώπων βρίσκονται σε ακραία φτώχεια και σε κίνδυνο τροφικής ε, ε, ε, φτώχειας. 20 εκατομμύρια από αυτούς είναι παιδιά και ψάχνουν εδώ στην Ευρώπη, Ευρώπη τα σκουπίδια για να βρουν το φαγητό που δεν μπορούν να έχουν σπίτι τους. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο, ε, να γίνεται μάλλον όλη αυτή η ιστορία για λίγα εκατομμύρια ευρώ για το 2012 και το 2013. Η φτώχεια χρειάζεται να αντιμετωπιστεί με βαθιά ε, μέτρα και όχι με πολιτικές λιτότητας που επιδεινώνουν τη φτώχεια και την ε, κοινωνικό αποκλεισμό. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη 4 η Ιουλίου συμπεριλαμβανομένη τη προώθηση μια συμφωνία για το ελάχιστο εισόδημα με τη βάση το 60% της μέσου όρου των ε, εθνικών εισοδημάτων. Θα θέλαμε λοιπόν να επιβάλλετε και πρόταση για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε. Ήλτα, για δύο λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως είναι αρμοδιότητα του δημόσιου τομέα να βοηθάει τους στοχούς. Και οπωσδήποτε οι πολίτες μας θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν να φάνε. Και βεβαίως... Γι' αυτό όλοι είναι υπέρ αυτού του προγράμματος. Να σας πενθυμίσω πως εδώ πέρα εγκρίναμε πρόσφατα την Ατζέντα 2020 και είπαμε πως στόχος είναι μεταξύ άλλων η καταπολέμηση της στόχιας. Τώρα λοιπόν να καταργούμε αυτό το πρόγραμμα δεν δείχνει και πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια. Ακόμα και αν γίνουν ακριβότερα τα τρόφιμα τα επόμενα χρόνια. Αλλά θεωρώ πως το πρόγραμμα αυτό δεν ξέρουμε αν είναι πράγματι, αν έχει στόχο να έχει την καταπολέμηση της φτώχειας. Δεν θα έπρεπε να είναι ο στόχος του, όπως ήδη ε, αναφέρθηκε στις ΙΠΑ ε, παραδείγματος χάρη, ότι είναι ένα ζήτημα και ένα μέσο γεωργικής πολιτικής για να μειωθούν τα αποθέματα και χρησιμοποιούν σημαντικό ποσοστό ε, η ΕΠΑ του προϋπολογισμού τους για τη Γεωργία ακριβώς για αυτό το σκοπό. Βεβαίως εμείς λειτουργούμε τελείως ε, διαφορετικά. Και πάντα ανοίγουμε το πρόγραμμα βραχυπρόθεσμα και διαπιστώνουμε πως είμαστε εντός του ιδίου δημοσιονομικού πλαισίου. Μακροπρόθεσμα όμως πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την απόφαση του ΔΕΚ και πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τον ίδιο στόχο με άλλα μέσα. Ένα λεπτό τώρα. Η κυρία Γκριλία. Κύριε Πρόεδρε, το Συμβουλίο Γεωργίας απέτυχε να προχωρήσει στην έγκριση αυτού του προγράμματο. Μιλάμε για 75% το οποίο πέρασε. Άρα χρειάζεται κατανόηση και να σταματήσουμε πρωτεύον την κοινωνία γιατί έχουμε τις, τους εθελοντές, έχουμε τις εθελοντικές οργανώσεις ε, που τώρα έχουν φυγεί. αυτό αμαυρώνει την εικόνα της Ένωσης, θα πρέπει να μπορέσουμε να πείσουμε τις αγορές όπως πήγες μπορώ σήμερα το πρωί, θα πρέπει επίσης τους πιο μη, μη προμήχους, αυτούς χρειάζεται να τους βοηθήσουμε, ε, αλλιώς πρόκειται για αδικία ε, αυτό θα κάνει μια κατάσταση κοινωνία εκρηκτική και όπως το είπατε κύριε Επίτροπε θα πρέπει και η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη αλλά και η Γαλλία να σταματήσουν τα κροκοδίλια δάκρυα και να συμφωνήσουν. Το είπατε κύριε Πρόεδρε είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Εάν το θέλουν την Δευτέρα θα κλείσει αυτό το θέμα ε, στην, στο, Συμβούλιο Απασχόληση Κοινών και Αποθέσεων. Θα πρέπει αυτό να γίνει ε, από, από αλληλεγγύη και σεβασμό προς αυτούς που το χρειάζονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ και κυρία και τώρα η κυρία Ντέσσαρνέζη έχει το λόγο για ένα μισή λεπτό. Το είδαμε με την κρίση του ευρώ, το είδαμε τώρα και με την υπόθεση αυτή των ε, τροφίμων ότι οι εθνικοί εγωισμοί έχουν ξαναγυρίσει δυστυχώ. Έχουμε τώρα αναδίπλωση και σωστρέφεια απλώς των κρατών μελών γιατί βλέπουμε ότι η αλληλεγγύη, το κοινοτικό πνεύμα ε, έχει τεθεί σε αμφισβήτηση αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Τώρα θίγονται οι πιο φτωχοί, αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν πιο μεγάλε δυσκολίε, εκείνοι οι οποίοι χρειάζονται περισσότερο αυτή την διατροφική βοήθεια από τι φιλανθρωπικέ οργανώσει. Έχουμε πάνω από 13 εκατομμύρια που το χρειάζεται αυτό στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν μπορεί, δεν πρέπει να του εγκαταλείψει, κύριε Επίτροπε, το είπατε και ο ίδιος με μεγάλη ακρίβεια το είπατε και το γράψατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει κάτι, να είναι παρούσα και θα πρέπει να σταματήσει αυτή την απαράδεκτη κατάσταση του μπλοκαρισμού στο Συμβούλιο. Είναι θέμα αξιοπρέπεια αυτών των λιγότερων προμοιούχο, ιδίω τώρα σε αυτή τη συγκυρία που μα έχει χτυπήσει η κρίση. Όμω, ε, ε, ακριβώ πρόκειται για την αξιοπρέπεια των ιδίων των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και οπότε πρόκειται για μια μάχη, για έναν αγώνα που σα το λέω, Επιτροπή και Συμβούλιο, ότι εμεί είμαστε στο πλευρό σα και όλοι εδώ ε, συσπηρωμένοι ε, στρατευμένοι σε αυτό το σκοπό. Ευχαριστώ ο πρόεδρος. ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντεσσαρνές και τώρα. Για ένα λεπτό. Πατρίκ Λεγιαρίκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πέρα από όλα τα ωραία λόγια που ακούγονται εδώ, υπάρχει ε, μια διπλή μαύρη κοιλίδα στο κούτελο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχήν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι διαπιστώντας διαρκώς την αύξηση της στόχης ως ένα φυσικό φαινόμενο. Πιστεύω πως αυτό σημαίνει την αποτυχία αυτής της υπερφιλελεύθερης Ευρώπης και η λιτότητα θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Έπειτα επίκειται επιζητιστική καταστροφή γιατί θέλουμε να διακόψουμε αυτή την επιζητιστική βοήθεια στους στόχους που αντίον θα έπρεπε να την αυξήσουμε. Μιλάμε για λιγότερο από 500 εκατομμύρια ευρώ για να επιτρέψουμε σε 18 εκατομμύρια ανθρώπους να τρώνε τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο μέρες. Ενώ έχει φτιαχτεί ένα πρόγραμμα για 440 δις για να εξασφαλιστούν οι τράπεζες. Σίγουρα υπάρχουν λιγότερε γεωργικέ παρεμβάσει όπω υπόθηκε, αλλά υπάρχουν, ξεκολουθούν να υπάρχουν επιδοτήσει για τι εξαγωγέ, κύριε Επίτροπε, άρα υπάρχουν χρήματα. Έπειτα μπορούμε να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο. Κοινωνική συνοχή για τη βοήθεια για του ε, πιο αδύναμου, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μειώνοντα τα κοινωνικά ταμεία και τα, το Ταμείο Συνοχή. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, Πατρίκ. Τώρα έχει δύο λεπτά ο συνάδελφο Μισελ Νταντά. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, εδώ και πάνω από τρία χρόνια η συζήτηση γύρω από το πρόγραμμα βοήθειας προς τους πιο αδύναμους βρίσκεται στην ουσία μπλοκαρισμένο στο Συμβούλιο. Αυτή η κατάσταση είναι παράδεκτη και είναι τόσο περισσότερο απαράδεκτη γιατί η εγκατάλειψη αυτού του προγράμματος ε, προβλέπεται για μια περίοδο που η Ήπειρός μας ε, ταλανίζεται από μια ανευπροηγουμένου κρίση. Ε, υπάρχουν ε, λοιπόν αυτοί που φτιάχνουν την Ευρώπη και οι άλλοι που την υπονομεύουν. Δεν πρέπει να καταστρέψουμε σήμερα αυτά που με υπομονή φτιάχτηκαν στο παρελθόν, ιδιαίτερα τη στιγμή που φαίνεται να να είναι πιο αδύναμος ο δεσμός ανάμεσα στα κράτη μας και που τα οθεί σε εθνικισμούς. Το να αποκατασταθεί το καθένα για τον εαυτό του ως μια αντίδραση, ένα αντανακλαστικό αποδεκτό, δεν αντιστοιχεί στην εικόνα μας για την Ευρώπη, ούτε στην εικόνα της χριστιανοδημοκρατίας στην οποία ανήκω. Ε, θα... Μια Ευρώπη που φτιάχνουμε εδώ και 50 χρόνια που δεν περιορίζεται σε μια απλή οικονομική συνεννόηση. Περιλαμβάνει αρχές που θα πρέπει, αξίες που θα πρέπει τώρα να αγκαλιάσουμε και πάλι και που τοποθετούν τον άνθρωπο στο επίκεντρο της πολιτικής. Ε, θα πρέπει να βγούμε από τις ε, στήρες ε, νομικές συζητήσεις για να λάβουμε τις δίκες και υπεύθυνε αποφάσεις. Κοινωνικό ταμείο μέσα στο πλαίσιο ενός ειδικού ταμείου και μέσα στο πλαίσιο της αναθεωρημένη ΚΑΠ, αν θα γίνει το ένα ή το άλλο, μα δεν είναι αυτό το ζήτημα. Η απόφαση του ΔΕΚ δημιουργεί μια επίγουσα κατάσταση που θα χτυπήσει 18 εκατομμύρια Ευρωπαίους που χαίρουν της επιστηστικής αυτής βοήθειας. Θέλω λοιπόν τώρα να αποφασίσουμε ποια είναι η κοινή μας εικόνα για την Ευρώπη και το μελλοντικό μας όραμα. Αυτό το θέμα δεν θα πρέπει καθόλου να περάσει από μια επανεθνικοποίηση μερική ή πλήρη της επιστηστικής βοήθειας. Μόνο και από κοινού θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα τεράστιε τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας. Μόνο κοινού θα μπορέσουμε να φανούμε ενωμένοι και αλληλέγγυοι και μόνο έτσι η πυρό μα θα μπορέσει αύριο να εξασφαλίσει έναν ορίζοντα ευημερία για το σύνολο των πολιτών τη. Κύριε Επίτροπε, εσεί προτείνατε μέτρα πολύ θαραλέα. Ο πρόεδρο διακόπτει τον ομιλητή. Σα τέλειωσε ο χρόνο. Έχει τελειώσει ο χρόνο σα, κύριε Νταντέν. Για ένα λεπτό ο κύριος Μάρκ Ταραμπέλα έχει τώρα το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Ε, εδώ δεν πρόκειται για συζήτηση. Πρόκειται για μια σειρά μονολόγων που κατευθύνονται στην ίδια κατεύθυνση, γιατί όλοι έχουμε την ίδια άποψη με κάποιε μικροδιαφορέ όσον αφορά τη διαδικασία. Αλλά πρέπει να επαναλάβουμε, δεν φταίει η Ευρώπη. Οι έξι κυβερνήσει των χωρών που ήδη αναφέρθηκαν πρέπει να τι επαναλάβουμε. Γερμανία, Αγγλία, Ολλανδία, Τσεχία, Δανία και Σουηδία χώρες επιπλέον που δεν είναι και από τις στοχότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι από τις πιο εγωιστικές ή που γίνονται σιγά σιγά πιο εγωιστικές. Πρέπει να καταλάβουν λοιπόν αυτές οι χώρες ότι οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Να... Αυτό, οδυναμία. αυτό που θέλω να κάνουν δύναμη με την... Ε, ε με το να μην βοηθήσεις κάποιον ο οποίος κινδυνεύει. Ιδιαίτερα για το 2012 και το 2013 που είναι μεταβατικές περίοδου πρέπει να φύγουν τα χρήματα από τη Γεωργία να μπουν στο κοινωνικό ταμείο και δεν θα πρέπει να το στερηθούμε αυτό. Βεβαίως ε, τα κράτη-μέλη είναι συνυπεύθυνα αλλά θα πρέπει η Ευρώπη να ντροπιαστεί σε αυτό το τόσο σημαντικό κοινωνικό θέμα. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Γκρίσμπεκ για ένα λεπτό. Πραγματικά μένω άναυδη όταν βλέπω τον Επίτροπο την Πολωνική Προεδρία και το σύνολο των συναδέλφων, όποιο και αν είναι τα έδρανα στα οποία βρίσκονται, ε, να έχουμε όλη την ίδια άποψη για τον σκανδαλώδη και να αξιοπρεπή χαρακτήρα αυτής της συζήτησης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βοήθειας στους πιο αδύναμους. Η απόφαση αυτή είναι σκανδαλώδης. Αυτή η αμφισβήτηση είναι ανεύθυνη από πλευράς των έξι κρατών που μπλοκάρουν ε, ή που θα μπορούσαμε να πούμε που ξεμπλοκάρουν, μάλλον που τα έχουν χάσει και που κινδυνεύουν να παίξουν μοιραίο ρόλο για αυτό που προσπαθούμε εμείς να φτιάξουμε. Όπως το είπε και ο Μάρκα, εγώ θέλω να καλέσω τους συναδέλφους που είναι σήμερα όλοι σύμφωνοι τους ε, Γερμανούς, Άγγλους, ε, Σουηδούς, Δανούς, Ολλανδούς και Τσέχους ε, συνάδελφους να ζητήσουν από τα κράτη τους να ασκήσουν πιέσεις στις κυβερνήσεις τους ώστε να πάψουν να κρατούν αυτή την αναξιοπρεπή στάση, αναξιοπρεπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το πολιτικό μήνυμα που μπορεί να είναι μοιραίο. Ευχαριστώ και συνάδελφε για τώρα. Για δύο λεπτά έχει το λόγο η κυρία Ράντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Μπαρόσο, αυτό το θέμα ε, το εξέθεσε στα πλαίσια των όσων είπε για την κατάσταση της Ένωσης ε, ελπίδα και ελληνική θα πρέπει να υπάρχει μέσα σε αυτή τη συγκυρία της κρίσης στην οποία είμαστε βυθισμένοι και γιατί όλο ένα και περισσότεροι βυθίζονται προς το κατόφλι της ε, φτώχειας. Θα πρέπει επομένως να, να πούμε ότι οι χώρες αυτές που αντιτίθενται σε αυτό το πρόγραμμα είναι το αντίθετο της αλληλεγγύης, θέτουν εις κίνδυνο την συνέχιση του, του, του, του προγράμματος αυτού με 1% του προπολογισμού ε, της Γεωργίας βοηθά 18 εκατομμύρια ανθρώπους. Ο, θα πρέπει να αποκαλύψουμε ποιοι είναι αυτοί. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι ανήκαν να δείξουν σήμερα ε, αλληλεγγύη. Παρακαλώ η, η Πολωνική Προεδρία να συνεχίσει προσπάθειες πριν τελειώσει τώρα η Προεδρία να καταφέρει τη συνέχιση προγράμματος γιατί αξίζει και, και το αξίζουν και, και εκείνοι που είναι επιλέξιμοι για να ωφελούνται και αποτελεί για ένα πάρα πολύ θετικό μήνυμα για τους πολίτες. Θα πρέπει το Συμβούλιο να λάβει υπόψη και την άποψη του Κοινοβουλίου, να συνεχίσει το πρόγραμμα και να βελτιωθεί έχει ζητήσει αυτό εδώ το σώμα. Να υποθυμίσω στους Αγίους και Κυβέρνησης ότι ελπίζουμε, ότι πιστεύουμε ότι στην επόμενη σύνοδο κορυφής θα δοθεί απεμπλοκή στο θέμα αυτό. Ε, ευχαριστούμε λέει ο πρόεδρος. Για άλλη μια φορά, κυρία μου, δεν μπόρεσαν οι διερμηνείς να παρακολουθήσουν το ρυθμό με την ταχύτητα με την οποία μιλάτε. Είπαμε ότι αντί να το λέει ο πρόεδρος υπάρχει ένα κουμπάκι στις κονσόλες και κάτι ανάβει ένα φωτάκι που σας λέει ότι έτσι όπως τα λέτε δεν μεταφράζεστε, το λέμε για άλλη μια φορά να το λάβετε υπόψη. Όταν ανάβει αυτό το φωτάκι στο μικρόφωνο πάει να πει ότι δεν είναι δυνατόν να μεταφραστούν αυτά που λέτε όπως τα λέτε. Το είπαμε και το ξαναείπαμε, δεν σας το λέω τώρα για να γνωρίζετε όλο τον μηχανισμό. Ναι, ναι, έχετε το λόγο για άλλη μια φορά. Δεν το ήξερα πρόεδρε ότι υπάρχει τέτοιο σύστημα. Μπορείτε να μου πείτε πού είναι αυτό το φωτάκι. Το έχω πει 25 φορές. Το λέω κάθε φορά που προεδρεύω για να το κάνουν και οι συνάδελφοι εδώ που προεδρεύουν. Ότι παίρνω εγώ αυτό το σινιάλο, ας το πούμε, από τους διερμηνείς. Σο, SOS λένε, κίνδυνος. SOS, οπότε και εγώ ε, το, το μεταφέρω στον ε, αγο, αγορητή, ούτως ώστε να επιβραδύνει και στη να πετάω εγώ το κουμπάκι και κάτι ανάβει στον οθόνη μπροστά σας. Κοιτάξτε, κοιτάξτε τώρα. Σβήνω το μικρόφωνο. Το σβήσατε εσείς. Ωραία. Βλέπετε μπροστά σας εκεί κάτι. Εκεί μπροστά. Α, συγγνώμη. Λέει η ομιλήτρια. Όμως, την ώρα που εμείς μιλάμε, είναι αδύνατο να δούμε τι, τι, τι, γίνεται στην, αυτό το αναβόσβησμα. Δεν το βλέπω. Αφήστε που γυαλίζει κιόλα. Ε, τότε να κάνουμε, κάνουμε ένα ηλεκτροσόκ, τι να κάνουμε, ένα, ένα κεραυνό, πώς θα γίνει. Ε, τι να κάνουμε, να, να, να, να χτυπάνε κάποια, κάποιο καμπανάκι. Καλά να δούμε όμως πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε. Έτσι, ένα καμπανάκι, ένα κουδούνι, το οποίο να χτυπάει, να χτυπάει και να το ακούει ο μιλητής. Τέλος πάντων, με την ευκαιρία σας το είπαμε. Η κυρία Γκαρθία τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Εράνθη Γκαρθία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικοστηρίου ξεκαθαρίζει το πόσο σημαντική είναι η συνέχιση του προγράμματος. Το είπαμε και στις δημοσιονομικές προοπτικές 14 έως 2020 σε σχέση με την επίτευξη του στόχου της μείωσης της φτώχειας. Να θα πρέπει να παραταθεί ο κανονισμός, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε ένα μηχανισμό, να συνεχίσει το πρόγραμμα και ο, προγραμμα... προγραμματισμός του προγράμματος σε σχέση με την κοινή πολιτική αυτά τα τρόφιμα να συνεχίσουν να καλύπτουν πάνω από 18 εκατομμύρια Ευρωπαίους που βρίσκονται σε κατάσταση ε, κοινωνικής περιθωριοποίησης. Θα πρέπει κάτι να γίνει με αυτή την παρεμποδίουσα μειοψηφία θέλουμε την αλληλεγγύη, γιατί θεωρούμε ότι είναι θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και βασικό το θεμελιώδες δικαίωμα, το δικαίωμα στην διατροφή. Αυτό το πρόγραμμα σήμερα παρά ποτέ χρειάζεται. Είναι θέμα συνείδησης, όχι χρημάτων. Κυρία Λεπάζου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, αγαπητοί μου συνάδελφοι. Η Ευρώπη δεν είναι μόνο μια νομισματική ή οικονομική ένωση. Οι συμπολίτε μας περιμένουν άλλα πράγματα, ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομική και κοινωνική κρίση. Κανένα δεν καταλάβει πω νομικοί λόγοι στερούν 18 εκατομμύρια άτομα από την τροφή. Πράγμα που είναι ένα θεμελιώδε δικαίωμα το οποίο αναγνωρίζουν οι συμβάσει μα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την ικανοποίησή μα και τη χαρά μα για τι προτάσει του, τα λόγια του Επιτρόπου και να ζητήσουμε από όλου να επιμείνουν να πιέσουν τι κυβερνήσει του ώστε το Συμβούλιο να πάρει την μόνη και μοναδική απόφαση που μπορεί να ληφθεί ε, ε, εφόσον υπάρχουν και τα κοινοτικά χρήματα να επιτρέψουν δηλαδή τη συνέχιση αυτής της βοήθειας την οποία να μπορούν να ζητήσουν με αξιοπρεπή τρόπο οι συμπολίτες. Με ένα θέμα αξιοπρέπειας και αλληλεγγύης. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Λεπάζ, το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Νικουλέσκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε πρώτα απ' όλα επιτρέψατε μου όπως ε, και οι συνάδελφοι να χαιρετήσω το ότι σήμερα ο κύριος Μπαρόζο αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα γιατί είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό το πρόγραμμα αυτό βοηθάει 18 εκατομμύρια Ευρωπαίους, δηλαδή πάνω από έναν στους 30. Ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση παλεύει με την κρίση και η φτώχεια υπάρχει παντού. Ο αγώνας κατά του αποκλεισμού είναι πάρα πολύ σημαντικός, πόσο μάλλον η επάρκεια των τροφίμων. Σήμερα είπε ο κύριος Μπαρόζο πως θα πρέπει να κάνουν τα θεσμικά όργανα αυτό το οποίο είναι αναγκαίο. Είμαι πεπισμένος πως θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες λύσεις για να βγούμε από αυτή την ε, κατάσταση. Τώρα, για τις δαπάνες αυτές και για την σπατάλη κάθε πολίτης ε, οι πολίτες συνολικά πετάνε 180 εκατομμύρια τόνους τρόφιμα κάθε χρόνος. Όμως η κατάσταση αυτή είναι απίστευτη και θα πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ρόντουστ κατόπιν. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Να πω κάτι, να ξεκαθαρίσει ευθύς εξ αρχής. Ως σοσιαλδημοκράτης εγώ θέλω να βοηθάω τους ανθρώπους ε, αυτό όμως σημαίνει να δημιουργηθούν θέσει εργασία για να έχουν οι άνθρωποι τη δυνατότητα να τραφούν μόνοι του. Κατά την άποψή μου, το πρόγραμμα αυτό, στην τωρινή του μορφή, δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Για μένα όλα αυτά είναι ελεημοσύνες και αναξιοπρεπή πράγματα. Και βεβαίως δεν είναι γεωργική πολιτική είναι κοινωνική πολιτική το να μοιράζουμε δωρεάν τρόφιμα και σύμφωνα με το δίκαιο το οποίο ισχύει είναι αυτό αρμοδιότητα των κρατών μελών. Υπάρχουν κάποια στήματα και στη Γερμανία που μοιράζουν ε, τρόφιμα από τα σούπερ μάρκετ. Σκεφτείτε, κάθε χρόνο πάνε 89 εκατομμύρια τόνοι τρόφιμα στα σκουπίδια. Είναι λογικό αυτό. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε λογικές ε, υποδομές για να μην εξαρτώνται οι άνθρωποι από ε, ελεημοσύνη. Και αυτό σημαίνει εξαρτησία με καλή δουλειά και καλές συντάξεις. Σας ευχαριστώ, κύριος Παπαστάμκος. Παρέλκει η επιχειρηματολογία υπέρ του αυτονοήτου. Η ανάγκη συνέχισης του επιστητικού προγράμματος υπέρ των απόρων, ιδίως υπό την τρέχουσα δυσμενέστατη κοινωνική συγκυρία, είναι επιτακτική. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να γίνει δεκτή η προτινόμενη δραστική μείωση των πόρων για το 2012. Ζητούμε άμεσα νέο νομικό πλαίσιο για την πλήρη αξιοποίηση των διαθυσίμων πόρων στο πλαίσιο της τρέχουσας δημοσιονομικής περίοδου καθώς και συνέχιση του προγράμματος κατά την μετά το 2013 περίοδο. Πέραν της αναγκαιότητας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων από τη δημόσια αποθυματοποίηση αλλά και από την αγορά, επιπλέον η επιλογή των διανεμωμένων προϊόντων οφείλει να μην περιορίζεται σε αυτά για τα οποία υπάρχει παρέμβαση αλλά να παρέχεται η ευχέρεια ευρύτερης επιλογής σε κάθε κράτος μέλος βάσει των πραγματικών αναγκών. η επιτροπή εισηγείται κύριε επίτροπε την καθιέρωση χρηματοδότησης. αντιλαμβάνεστε βεβαίως τη δυσκολία αν όχι την αδυναμία που συνεπάγεται η πρόταση αυτή για ορισμένα κράτη μέλη τα οποία έχουν μεγαλύτερη ανάγκη χρήση του προγράμματος. τέλος σε όσους ζητούν επανεθνικοποίηση των επισυτιστικών προγραμμάτων ως υπόθεση κοινωνικής πολιτικής εκάστου κράτους μέλους απαντώ ότι πέραν της κοινωνικής του διάστασης το πρόγραμμα συμβάλλει στην σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών και του γεωργικού εισοδήματος στην ένωση. πολλό δε μάλλον σηματοδοτεί συμβολισμό ελάχιστης έκφρασης αλληλεγγύης υπέρ των απόρων πολιτών τη. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπερές, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Βόντα του Συμβουλίου, αυτή η υπόθεση δεν είναι υπόθεση επικουρικότητας, διότι η κοινωνική βοήθεια και ο αγώνας κατά τις στόχες είναι υπόθεση όλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι υπόθεση επικουρική παράπλευρη, είναι μεγάλη υπόθεση. Επιτρέπει σε ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση μεγάλης φτώχειας, μεγάλης ένδυας, να μην ζητιανέψουν, αλλά να μπορέσουν να τραφούν. Κανένα δεν μπορεί να αποφύγει να στρέψει την προσοχή του από αυτού τους στόχους. Ο πρόεδρος της ε, Κοινοκομισιόν σήμερα το πρωί μας είπε ότι είναι πλέον καιρός ο χρηματοπιστωτικός τομέας να πληρώσει τη ζημιά αυτής της κρίσης. Και το λέμε και εμείς ότι είναι καιρός ο υπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσει να βοηθά το του έργο που κάνουν αυτοί που λειτουργούν ε, τις τράπεζες τροφίμων και επιτρέπουν στους ανθρώπους που βρίσκονται στην, ε, σε ακραία φτώχεια να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάποια στοιχεία δεν θα δεχτούμε όμως ούτε να οργανώνεται η αλληλεγγύη των φτωχών με τους φτωχούς. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να χρηματοδοτηθεί και σίγουρα θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί υπό το τίτλο της κοινωνικής βοήθειας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει να υπάρξει αντιστάθμιση. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, εμείς σας το λέμε, κάνετε ό,τι μπορείτε ε, χρησιμοποιήστε κάθε δυνατότητα ώστε να λυθεί από τη Δευτέρα και αυτή η υπόθεση γιατί θα κριθείτε στον απολογισμό της Προεδρίας σας. Σας ευχαριστώ κυρία Νέντελ Τσέβα είναι η επόμενη. Αγαπητοί συνάδελφοι, κανένας ανάμεσά μας δεν, παραμένει ασυγκίνητος στο γεγονό ότι 40 εκατομμύρια Ευρωπαίοι απειλούνται από τη φτώχεια και ότι 13 εκατομμύρια εξαρτώνται από αυτό το πρόγραμμα το επισητιστικό και το χειρότερο είναι ότι αυτή η κατάσταση θα ε, επιδεινωθεί. Θα και να μπορέσει να σεχθεί αυτό το πρόγραμμα γιατί αυτού του είδους η μεγάλη περικοπή που έχει γίνει πρόκειται να ε, προλάβει το πρόγραμμα αυτό και σήμερα και αύριο και θα πρέπει επομένω να διανεμηθούν θα τα σε αυτού που το χρειάζονται, τόσο ώστε να σταματήσει η εξάρτησή τους. Όμως ε, θα πρέπει να τους δώσουμε μια ευκαιρία, ούτως ώστε ε, αυτοί οι άνθρωποι να, να, προχωρήσουν. Οπότε έχουμε τώρα τα ιδιωτικά ταμεία που είναι πάρα πολύ σημαντικά. παρόλα αυτά όμως χρειάζεται υγιεινή διατροφή που είναι κάτι πάρα πολύ βασικό από την παιδική ηλικία και μετά. Άρα ο δικό μας ρόλο είναι να βοηθήσουμε αυτόν τον κόσμο και έτσι να σταματήσει να ε, να να, οι άνθρωποι να εξαρτώνται αυτό το πρόγραμμα γιατί δεν μπορούν να συνεχίζουν. Οπότε τα προγράμματα, τα προ... οι προτάσεις που μου γίνει σημαντικές και οπότε η καταπολέμηση της φτώχειας είναι ένας ε, στόχος για τις χιλιετίας άρα χρειάζεται μια τέτοια πολιτική για τα ίδια διατροφής ούτως ώστε να σταματήσει αυτό το είδος εξάρτηση και να μην ξεχνούμε τις βασικές μας αρχές, να μην ξεχνούμε τις υποθέσεις που έχουμε δώσει. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, κυρία Ντάντζελα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, το Ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα εξητιστικής βοήθειας ε, θα συνεισφέρει στην ενίσχυση και της κοινωνικής πτυχής πέρα από την κυριαρχική πολιτική. Βοηθάει ανθρώπους που είναι φτωχοί, ειδικά στα πλαίσια της ε, τόλμης κρίσης. Θεωρώ αναγκαίο τα άτομα τα οποία χρειάζονται βοήθεια να συνεχίσουμε να τα υποστηρίζουμε στο επίπεδο του τρέχοντος έτους. Ξέρουμε πως έχει και κοινωνική πτυχή αυτή η πολιτική. Λόγω λοιπόν της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης ε, θα πρέπει να αναγνωρίσουν τα έξι κράτη-μέλη που αναφέρθηκαν την κατάσταση και να βοηθήσουν στον περιορισμό της φτώχειας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ η κυρία Μωρέν Σαρτιέ. Ευχαριστώ. Έχουμε το καθήκον να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για αυτό που έχει πλήξει ε, του, τους πιο αδύναμους και ε, ακριβώς μας αφορά πάρα πολύ και θέλουμε να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα που αποτελεί έκφραση κοινοτικής ελληνικής. Τρία είναι τα μηνύματα. Πρώτα-πρώτα προς την Προεδρία του Συμβουλίου να δούμε ε, κατά πόσον θα, θα, θα, αποδείξει το Συμβούλιο ότι σέβεται τις βασικές ε, αρχές της ε, κοινότητας και να σταματήσει αυτούς οι οποίοι αποτελούν παραδείγματος ψηφία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να δούμε τι θα γίνει με την πρότασή σας κύριε Πρόεδρε που θέλετε το πρόγραμμα αυτό να ενταχθεί στο κοινωνικό ταμείο το οποίο όμως είναι το πρώτο μέσο πολιτικής για την κοινωνική ένταξη μέσω της ε, επαγγελματική ένταξης οπότε και θα πρέπει το πρόγραμμα ακριβώς όπως έχει να συνεχιστεί όχι να βελτιωθεί και να συνεχίσουν να δίνονται τα τρόφιμα σε αυτούς που έχουν ανάγκη και αυτό θα μας έχει σε ε, κινητοποίηση. Όλοι εδώ έχουμε κινητοποιηθεί. Το μήνυμα το τρίτο είναι προς τους βουλευτές ε, εκείνους από τις χώρες της εμπλέκουσας, της παρεμπιδούσας μειοψηφίας θα πρέπει από σήμερα να δώσουν το μήνυμα στις κυβερνήσεις τους και το μήνυμα είναι ότι θα πρέπει να πάψει αυτή η θλιβερή ε, θέση τους η οποία μπλοκάρει την Ευρώπη. Πρόεδρος. Τώρα έχουμε τη διαδικασία κάτσε Πάρα πολλοί ζητούν το λόγο. Δεν μπορείτε να καλυφθείτε όλοι. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ. Και αντίστοιχα με ο πρώτος. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ναι, γίνεται λόγο για του φτωχού για την αλληλεγγύη. Και στο Συμβούλιο Γεωργίας έχουμε περιποδίου σε μια ψηφία η οποία δεν θέλει να τοποθετεί αυτό ο κανονισμός τόσο ώστε να ρυθμιστεί το θέμα ενίσχυση ενίσχυσης της αρρωγής με, μέσω τροφίμων το, το, το μήνυμα το πήρε ο κ. Σαβίτσκι, όμως θα πρέπει να δείτε το 60% της πρικοδότησης χρειάζονται ούτως ώστε 79 ε, εκατομμύρια κόσμο να μπορέσουν να, να, να, να γιατί αυτοί ζουν κοντά στο κατόφλι φτώχειας ή κάτω από αυτό. Όλα αυτά ε, τα δίνουν οι κυβερνήσεις, οι αρχές, οι τοπικές, οι περιφερειακές, οι μη κυβερνήσεις οργανώσεις. Η δευρωμαϊκή Ένωση ε, συγχρηματοδοτούσε κατά 40%. Η θέση αυτών που παρεμποδίζουν ως μειοψηφία ε, δημιουργεί πρόβλημα για του χρόνου και απειλεί με εξαφάνιση το πρόγραμμα το 2013 καταδικάζουν τη θέση τους Και ευχαριστούμε την Πολωνική Πρωτεία, ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δείχνουν αποφασιστικότητα ώστε να διτηρηθεί το πρόγραμμα. Επίση, ε, κατηγορηματικά καταδικάζουμε τη θέση αυτών των παρεμποδιζουσών χωρών και του λέω, του ρωτώ, πού πήγε η, η, η ανθρωπιά τους Κύριε Τσόλος, ε, κουράγιο, διότι κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να αντιταχθεί στην ανθρωπιά ή στον ε, νόμο του Θεού. παρακαλώ να, ανατηρεί τα χρονικά ωραία, λέει ο Πρόεδρος, γιατί τελείω δεν μπορούσαν οι συνάδελφοι να, να λάβουν το λόγο. Η κυρία Κάλμπαχ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Κύριε Υπουργέ, συζητήσαμε σήμερα την κατάσταση της Ένωσης και μιλάμε και για αλληλεγγύη και πόσο κοινικά ακούγονται αυτά τα λόγια στους Ευρωπαίους όταν ε, τους λέμε «Α, δεν έχει ξεκαθαρίσει η νομική κατάσταση, οπότε πεινάστε εσείς μέχρι να τα βρούμε». Δεν είναι δυνατόν, δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία καθυστέρηση αν υπάρχουν άλλες νομικές λύσεις, αυτές είναι για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή χρειάζον, χρειαζόμαστε τρόφιμα για αυτούς που δεν έχουν να φάνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μποβέ. Euh, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εγώ δεν θα επαναλάβω τόσα ήδη υπόθηκαν, αλλά πιστεύω πως υπάρχει όντως ένα πραγματικό πρόβλημα αξιοπιστία για την Ευρώπη σήμερα, μετά όσα συμβαίνουν. Ε, κάνουμε μια νομική διαδικασία που μας λέει από μια πλευρά υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική και από την άλλη οι πολιτικές των κρατών. Αλλά όταν το 58 η συνθήκη της Ρώμης μας λέει ότι το να εγγυηθούμε την διατροφή όλων των Ευρωπαίων και την ε, τροφική ασφάλεια, είμαστε μέσα σε μια ευρωπαϊκή πολιτική και όχι σε πολιτική των κρατών. Σήμερα αυτό που δείχνει αυτή η κατάσταση, πέρα από τον εγωισμό ορισμένων κρατών, είναι ότι δεν ε, ε, ε, είναι πως δεν έχουμε αρκετή Ευρώπη, αλλά δεν έχουμε αρκετή ευρωπαϊκή βούληση από ορισμένου αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων. Γι' αυτό και θέλω να χαιρετήσω τον Ευρωπαίο Επίτροπο κ. Σιόλο, που σήμερα μιλά στην εφημερίδα Le που είχε και το, η παρεσία να αναγνωρίσει πω αυτή η πολιτική είναι απαραίτητη για του πιο φτωχού Ευρωπαίου. Αν δεν είμαστε σε θέση να αμφισβητήσουμε την απόφαση του Συμβουλίου, αυτή η Ευρώπη θα. Ε, ε, αποχαρακτηριστεί από τους πολίτες. Ευχαριστώ κυρία Μαγκίνες. Κύριε Πρόεδρε, το μήνυμα του Κοινοβουλίου είναι σαφές, θέλουμε να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα λόγω της ανθρωπιστικής του πτυχής. Άκουσα την συζήτηση και αναρωτιόμουν αυτοί οι οποίοι επωφελούνται από αυτό το ζήτημα ασχολούνται με τη νομική βάση, βάση την οποία τους μοιράζουν φαΐ ανησυχούν για τις λεπτομέρειες που μας απασχολούν εμάς εδώ πέρα. Υπάρχουν πολλοί έξυπνοι άνθρωποι εδώ πέρα για να βρουν μια λύση. Δεν θέλω να καταδικάσω τα κράτη-μέλη που μπλοκάρουν εδώ πέρα. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Θέλω να προσπαθήσω να τους πείσω για την αξία αυτού του προγράμματος για την αλληλεγγύη της Ένωσης. Θέλω μια βραχυπρόθεσμη λύση για τα επόμενα δύο έτη, αλλά όπως είπε και ο Τζιμ Νίκολσον, θα ήθελα να ξαναδούμε το τι θα κάνουμε μετά το 2014. Καμιά φορά πρέπει να γίνουν τα πράγματα διαφορετικά, αλλά τώρα υπάρχει άμεσο πρόβλημα στην Ιρλανδία. Υπάρχει ένα εκατομμύριο ευρώ το οποίο θα χαθεί από αυτή τη βοήθεια, οπότε χρειάζεται μια άμεση λύση. Και απευθύνω έκκληση να μην μπλοκάρουν αυτοί που μπλοκάρουν. Ευχαριστώ κύριο Στέρκας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Και εγώ συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους που το είπαμε και στις 4 Ιουλίου ότι θέλουμε να σας βοηθήσουμε και θα πρέπει να αρθεί αυτή η μεγάλη ντροπή. Είναι κατανόητο αυτό που κάνουν αυτές οι πέντε χώρες στο Συμβούλιο. Δεν είναι δυνατόν να σταματάνε την πρόοδο της κοινοτικής αλληλεγγύης. Μην ξεγελιόμαστε έτσι. Δεν καταπολεμούμε την ε, φτώχεια που έχουμε 80 εκατομμύρια φτώχους αλλά έχουμε αυτά τα 13 εκατομμύρια που πεινάνε, την πείνα καταπολεμούμε. Κάντε περικοπές όπου θέλετε, αλλά προς Θεού όχι για αυτό το πρόγραμμα. Παρακαλώ, αλλάξτε τη γνώμη του Συμβουλίου. Θέλω να μάθει όλος ο κόσμος ότι εμείς οι βουλευτές θέλουμε να άρουμε αυτή την ντροπή. Επομένως, να βρεθεί κάποια λύση για αυτούς που είναι πιο, ε, αυτοί που έχουν πιο, πιο μεγάλη ανάγκη, που είναι μη προνομιούχοι. Σταματήστε την ντροπή, γιατί πρόκειται για μια ε, Ευρώπη που ξοδεύει τα λεφτά, μια Ευρώπη του, του, του πλούτου, που πρέπει να δείξει ελληνική. Ευχαριστώ. Μαύρο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να βοηθήσω να αποσαφινιστεί ένα παράδοξο. Η αρχή της επικουρικότητας ε, όχι μόνο υπερασπίζεται τι αρμοδιότητες των κρατών, αλλά αναφέρεται σαφώ και στο γεγονός ότι αν κάποιο κράτος δεν είναι ικανό να νομοθετήσει, παρεμβαίνει το ανώτερο επίπεδο ε, με επικουρικό τρόπο. Άρα λοιπόν είναι βάσιμη η δυνατότητα παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλά το κατάλαβε η Προεδρία της Πολωνίας αλλά και η Κομισιόν. Οφείλουμε λοιπόν σε αυτέ αυτές τις περιστάσεις να κινητοποιήσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να απαντήσουμε στην ανάγκη 18 εκατομμυρίων ανθρώπων των οποίων το κρατικό επίπεδο ε, ε, κάποιων κρατών δεν μπορούν να καλύψουν. Και πρέπει επίσης να προσέξουμε, δηλαδή Θέλουμε να, μεταφέρουμε, να μεταφέρουμε στην, στο κοινωνικό κεφάλαιο. Ωραία, αλλά προσοχή, θα χάσουμε την αρετή ε, το θετικό στοιχείο του γεωργικού κλάδου που μπόρεσε να διαχειριστεί τον μηχανισμό και δεν θα μπορούμε να αποσαφηνίσουμε οπότε η κοινωνική υπόθεση θα είναι εθνική αρμοδιότητας ή κοινοτικής αρμοδιότητας. Σας ευχαριστώ. Κυρία Κρέτσου. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα συμφωνήσω και εγώ με όσου μίλησαν για εγωισμό των έξι κρατών μελών που μπλοκάρουν. Πέρσι είχαμε το έτος καταπολέμησης της στόχιας. Αλλά μόνο λόγια. Γιατί εάν είναι να δούμε τι γίνεται στην πράξη, οι κυβερνήσεις δεν δείχνουν αλληλεγγύη. Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα από τα λίγα μέσα με τα οποία βοηθά άμεσα τους πολίτες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πάνω από 40 εκατομμύρια άνθρωποι που είναι φτωχοί, γι' αυτό θεωρώ πως η μη επιμήκυνση αυτού του προγράμματος είναι κάτι το πολύ δυσάρεστο. Θεωρώ πως το πρόβλημα της χρηματοδότησης από τον προπολογισμό της Γεωργίας είναι μια δυνατότητα και θα πρέπει η λύση να βρεθεί στο μότρο δυνατόν. Ευχαριστώ τελευταίος ο μιλητής κυρία Ντεβό. Έξι κράτη-μέλη κρατούν στα χέρια τους την τύχη 18 εκατομμυρίων Ευρωπαίων που χρειάζονται βοήθεια. Αυτά τα έξι κράτη-μέλη έχουν γίνει δικαστές, αλλά άλλο δικαστής, άλλο ανθρωπιστής. Επομένως θα πρέπει να εκφράσουμε θυμό σε αυτούς οι οποίοι κοφεύουν στα σήματα κινδύνου όλων που ζητούν να βοηθήσουμε τους πιο αδύνατους. Και εμείς τώρα που είμαστε οι βουλευτές που εκπροσωπούμε όλους τους Ευρωπαίους να βάλουμε στην άκρη τους εθνικιστικούς ε, ε, εγωισμούς και θα πρέπει να βοηθήσουμε, είπαμε, και εκείνους τους, Ευρωπαίου Ευρωπαίους των, χωρών που έχουν οικονομικά προβλήματα και άρα θα πρέπει τώρα να δούμε ένα θέμα η νομική βάση, αλλά επίσης άμεσα να, να, να μην σταματήσει αυτό το πρόγραμμα το 2012 μέσα σε αυτή την τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία της κρίσης. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, και τώρα θα δώσουμε τον ε, λόγο στον Επίτροπο για να συνοψίσει αυτά της συζήτησης και να απαντήσει αν θέλει στους ερωτήσεις έχουν ε, εγώ θα ήθελα ο κύριος Τσόλος να προβώ σε κάποιες ε, διευκρινήσεις για τις παρατηρήσει που κάποιοι από εσά έχουν διατυπώσει. Όχι, δεν θέλω να πείσω αυτούς που είναι ήδη πεπισμένοι για τη συνέχεια του προγράμματος. Ίσως θα πρέπει να δούμε με αυτή την ευκαιρία πώς θα ακουστεί αυτό το μας το μήνυμα εκεί που πρέπει να ακουστεί. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα κοινωνική πολιτική. Ε, το οποίο έχει σχέση και με εθνική αρμοδιότητα. Έχει επομένως Έχουμε πει ότι εμεί κάναμε την επιλογή μας για 2014-2020. προτείνουμε να προκοδοτηθεί αυτό το πρόγραμμα στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής και ε, κοινωνικής ένταξης. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Ε, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι εθνική αρμοδιότητα. Αυτό είναι ζήτημα πολιτικής απόφασης η πλειοψηφία νομίζω το αποφάσισε για την περίοδο 2014-2020. Τώρα όμω λέμε ότι έχουν τεθεί να αμφιβόλο το τι θα γίνει 2012-2013 ε, το Κοινοβούλιο όπως και το Συμβούλιο συμφωνήσατε για τον προπολογισμό ότι αυτό το πρόγραμμα θα ενταχθεί ε, στην κοινή πολιτική. Όμως είναι αλήθεια ότι άλλαξαν τα πράγματα και είπαμε ότι το σούτο μάλλον ισχύει ε, το, ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν θέτει ένα αφιβολία τον κανονισμό. Ίσα ίσα λέει ότι θα πρέπει να τηρείται ο εγκριθής ε, κανονισμός και η Κομισιόν αυτό θέλει. Ε, να συνεχίσει να τρέχει, να ισχύει ο, ο κανονισμός για να κάνουμε τη δουλειά μας. Όμως εμείς δεν κάνουμε πολιτική. Λέμε ότι θα πρέπει αυτοί που πρέπει να λάβουν την πολιτική απόφαση. Εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε και κατεβάσαμε την νομοθετική πρόταση ούτως ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε επίσης και το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο όμως δεν κόβει τις ε, αγορές, τις από την αγορά. Απλώ λέμε ότι, ε, ότι δεν μπορούμε τώρα Όπω ισχύει ο κανονισμό να πάμε στην αγορά να ψωνίσουμε, τότε α τροπήσουμε τον κανονισμό. Γι' αυτό φτιάχνει ο κανονισμό για να επιδέχεται μεταβολέ και τροποποιήσει. Τώρα, το ότι από το 2014 εντάσσεται στην κοινωνική πολιτική αυτό το πρόγραμμα δεν μας εμποδίζει τώρα να λάβουμε απόφαση ε, με μια κοινή ε, νομική βάση. Είπαμε ότι έχουμε 100 ε, εκατομμύρια ευρώ απόθεμα και έτσι μπορούμε να έχουμε την νομική βάση για την αγροτική πολιτική. Αυτό το οποίο προτείνει το Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να παραμείνει αυτή η διτή, η διπλή νομική βάση και αυτή που σχέση με την ΚΑΠ και αυτή που σχέση με την κοινωνική πολιτική. Θα κάνουμε την πρόταση στο αρμόδιο Συμβούλιο στην αρχή της επόμενης εβδομάδας και ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής ή το Συμβούλιο Γεωργίας θα καταφέρουν να λάβουν μια απόφαση. Είπατε και για την ε, συγχρηματοδότηση ότι κάποια κράτη-μέλη δεν μπορούν να, να συμφωνήσουμε τη συγχρηματοδότηση όπως είχαμε εμείς προτείνει. Ήδη επανειλημμένα σας είπα ότι πρώτη να αναθεωρήσουμε την, τη μέθοδο της συγχρηματοδότησης εάν αυτό εμποδίζει τη λήψη απόφασης και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να λάβουμε κάποια απόφαση είναι θέμα και δικό μας αλλά βέβαια και της Προεδρίας και εμείς και η Προεδρία είμαστε αποφασισμένοι ε, τώρα κύριε Νίκολσον έχουμε διασπάθηση χρημάτων και πρέπει να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τη λειτουργία του προγράμματος αλλά για την αποτελεσματικότητα έχουμε ένα πρόγραμμα το, για το οποίο έχουμε κάποια νούμερα 340 εκατομμύρια τόνους που ε, μοιράζονται σε 18 εκατομμύρια επιλεξίμων. άρα υπάρχουν επιλέξιμοι πίσω από αυτά τα χρήματα και σας βεβαιώ ότι αυτή η πόρια είναι 500 εκατομμύρια που έχουμε τώρα και χρησιμοποιούνται ως ε, μοχλός για την συλλογή κάποιων προϊόντων που δεν ε, διασπαθίζονται και έχουν και αυτές τις διατροφικές τράπεζες κάποια καταστήματα. Οπότε δίνονται όλα αυτά στους πιο αδύνατους και έτσι έχουμε αυτά τα προγράμματα βοή, αρρωγής. Άρα χρησιμοποιούνται αυτά τα, πιάνω τόπο αυτά τα χρήματα. Και τα 500 εκατομμύρια χρησιμοποιούνται ως μοχλός για να βρεθούν ακόμη πολύ περισσότερα χρήματα σε δύο κρατών μελών. Για μια φορά σας επαναλαμβάνω ότι ελπίζω, σχεδόν πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε ε, σε συνεργασία με το Συμβούλιο να πετύχουμε την κατάλληλη πλειοψηφία για να συνεχίσει να τρέχει το πρόγραμμα. Ε, ε, ακόμα δεν, δεν, δεν έχει περάσει ε, δεν έχουμε την τελευταία ευκαιρία, αλλά σε λίγο ε, ο χρόνος τελειώνει. Ευχαριστούμε πολύ, ο Πρόεδρος. Και τώρα τελευταίος, αλλά σημαντικός. Θα λέω το λόγο για το Συμβούλιο, ο κύριος Σαββίτσκι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Επίτροπε. Να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση αυτή οπωσδήποτε θα με βοηθήσει να κόψω τον γόρδιο δεσμό που υπάρχει από το 2008. Θα υπενθυμίζω πως έκτοτε έχουν περάσει έξι προεδρίες και αρχίζει γενομένης από τη Γαλλική Προεδρία κάθε Προεδρία πέρασε το θέμα αυτό στην επόμενη. Θα έλεγα λοιπόν πως η Πολωνική Προεδρία δεν θέλει να δώσει με τη σειρά της το πρόβλημα αυτό στον επόμενο. Θέλουμε να λυθεί το πρόβλημα άμεσα ως πολιτικός. Πρέπει να πω πως ντρέπομαι για το ότι η πλειοψηφία, η μειοψηφία η οποία μπλοκάρει αποτελείται από χώρες οι οποίες στο παρελθόν είχαν χρησιμοποιήσει πολύ τον μηχανισμό παρέμβασης στην αγορά και ποτέ δεν είχαν πρόβλημα με το να μοιράζονται τα αποθέματα του μηχανισμού στους στοχούς. Τώρα δημιουργούμε ένα τεχνητό νομικό πρόβλημα και μας είπε ο Επίτροπος δεν είναι πρόβλημα νομικό ή χρηματοδότησης αλλά πολιτικό εδώ σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εθετήσατε το εξαπλό πακέτο, ένα πακέτο διάσωσης για τις τράπεζες. Οι έξι αυτές κυβερνήσεις δεν τρέπονται. Όταν δεν λαμβάνεται μία απόφαση να βοηθήσουμε 18 εκατομμύρια ανθρώπους με ένα συγκριτικά μικρό ποσό. Χαίρομαι που είχαμε πολιτική συζήτηση και δεν κρύβουμε το κεφάλι μας στην άμμο. Πριν από μία εβδομάδα έθεσα το ζήτημα αυτό σε μία δημόσια συζήτηση του Συμβουλίου γιατί θέλω να μάθουν οι λαοί της Ευρώπης ποιος λέει τι και γιατί. Και τώρα, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ πως μετά από αυτή τη συζήτηση η συνείδηση των κυβερνήσεων εκείνων που μπλοκάρουν θα ε, πρέπει να έχει αφυπνιστεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σαβίτσκι. Εδώ πέρα τελείωσε η συζήτηση για αυτό το θέμα και περνάμε στο επόμενο θέμα.